θεμέλια στην εκπαίδευση για τη σημερινή οικονομία με ανταλλαγή ε, εμπειριών και με τα λεγόμενα ε, παλιά κράτη-μέλη, με τα νέα κράτη-μέλη συνεργάζονται καθημερινά στην Ευρώπη. Δύο ακόμα σχόλια. Δεν είναι καθόλου παροχημένα αυτά τα πράγματα και παλιωμοδίτικα. Είναι πάρα πολύ σύγχρονα και το ένα δισεκατομμύριο τώρα σχεδόν που απελευθερώνεται για την ε, εκτέλεση καινοτόμων προγραμμάτων είναι πολύ σημαντική. Πολλές φορές θέλει κάποιος να κάνει ένα πρόγραμμα κοντά στα σύνορα και ψάχνει συνεργασίες για να δημιουργήσει κλίμακα, ας πούμε, σε νέες τεχνολογίες, στην τρισδιάστατη εκτύπωση. Τώρα όμως ε, ε, χρειάζεται διαπεριφερειακή συνεργασία ε, ε, εδαφική συνεργασία ε, και δεν είναι αυτό καθόλου ξεπερασμένη πολιτική, είναι πάρα πολύ επίκαιρη και θα τα δούμε και στο επόμενο πλαίσιο και στο επόμενο πρόγραμμα. Και μπράβο σας. Πολύ συναρπαστικά αυτά που λέτε, αλλά τελείωσε ο χρόνος σας, λέει ο Πρόεδρος. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, η κυρία Μερσέτης Μπρέσο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Για τρίτη φορά, Πρόεδρε. Και εγώ, όπως και άλλοι, προέρχομαι από μία όμορη περιοχή. Γι' αυτό το Interreg ήταν ε, ένα πολύ καλό μέσο για τη συνεργασία περιφερειών. Και νομίζω ότι αυτό είναι μία προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όλα αυτά τα χρόνια, χάρη στο Interreg, προώθησε ένα πρότυπο ανάπτυξης και ειρήνης και πολλές τοπικές αρχές συνεργάστηκαν σε σχέδια που βελτίωσαν την ζωή των πολιτών. Επίσης αναπτύξαμε μέσα όπως το, ε, την Ευρωπαϊκή Ομάδα περιφερειακής συνεργασίας και ούτω καθεξής. Είμαστε υπερήφανοι γιατί ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη στιγμή επιτύχαμε να δώσουμε 11 δις ευρώ για την επόμενη θητεία επαυξάνοντας τα αποτελέσματα της Επιτροπής. Ελπίζουμε να επιβεβαιωθούν οι προσδοκίες μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Από τους φιλελευθέρους, ο κύριος Βαν Μίλτεμπερκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η διασυνορική συνεργασία είναι ε, από τις πιο ορατές εκφάνσεις της ευρωπαϊκής συνεργασίας. Τα προγράμματα Interreg εδώ και δεκαετίες ε, λειτουργούν σωστά προς την κατεύθυνση αυτή. Ο κόσμος πηγαίνει, έρχεται, δουλεύει από την άλλη πλευρά των συνόρων, ε, χρησιμοποιεί τις υποδομές. υπάρχουν καλύτερες διασυνδέσεις. Χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προωθεί αυτή την συνεργασία και οικονομικά. Και χρειάζονται χρήματα γιατί στο μέλλον ε, χρειάζεται ε, να χρηματοδοτηθούν, όπως ακούσαμε, οι καινοτόμες επενδύσεις. Περίπου ένα δισεκατομμύριο για κοινέ ε, επενδύσεις, ιδρύματα εκπαιδευτικά, επιχειρήσεις και σε διάφορα κράτη-μέλη της Ένωσης. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να αναπτύξουμε νέα προϊόντα, νέες υπηρεσίες και να τα βγάλουμε στην αγορά. Και αυτό που έχει σημασία δεν είναι που βρίσκεται η επένδυση, ε, αλλά αν έχει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για να έχει και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Σε ε, ευρωπαϊκή κλίμακα, αν επενδύσουμε σε ε, καινοτομία, μπορούμε παγκόσμια να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί απέναντι στις ΗΠΑ ή στην Κίνα. Με καλή συνεργασία, λοιπόν, και στην Ευρώπη δημιουργούμε και περισσότερη ε, εργασία, περισσότερες θέσεις εργασίας, περισσότερη ευημερία και περισσότερο πλούτο. Ελπίζω γρήγορα να αρχίσετε να διαπραγματεύεστε αυτό το νέο κανονισμό με το Συμβούλιο. Είναι σημαντικό τα νέα προγράμματα Interreg το 2021 να ε, αρχίσουν να λειτουργούν με ταχύς ρυθμούς και να ε, συνεχίσουν αυτό το ευεργετικό έργο σε όλη την Ευρώπη και σε όλες τις παραμεθορίες περιοχές. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ροπέ. αποουσιάζει μάλλον ο κύριος Τσέλε. Ευχαριστώ πολύ στα πολωνικά, κύριε Τσέλερ. Κύριε Επίτροπε. Είναι σημαντικό που η έκθεση αυτή συνοδεύεται από συζήτηση. Ακόμα και αν είναι άγρα μεσάνυχτα, αξίζει τον κόπο να το κάνουμε, γιατί στην αρχή είχε προβλεφθεί μόνο μια σύντομη παρουσίαση στην Ολομέλεια, χωρίς συζήτηση. Δεν υπάρχει σχεδόν κανένας άλλος τομέας ευρωπαϊκής πολιτικής που να ανταποκρίνεται τόσο πολύ ε, στη συνεργασία πέρα από σύνορα και στην ε, συνοχή της Ένωσης ε, και που να εγγράφεται σε αυτό το στόχο, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία. Ε, τα ευρωπαϊκά σύνορα έχουν γίνει όλο και περισσότερο περατά, αλλά παρά αυτά είναι διαφορετικές οι διοικητικές δομές και η ένωμη τάξη, ε, πράγμα που ε, δυσκολεύει τη διασυνοριακή συνεργασία και την κυκλοφορία γύρω στα σύνορα. Ε, σε αυτές τις περιφέρειες που δεν έχουν πολλές υποδομές βοηθούμε τους πολίτες να λύσουν από κοινού τα προβλήματά τους και να ελοποιήσουν τα προγράμματά τους. Για να συνεχιστεί η ε, ευρωπαϊκή αυτή εδαφική συνεργασία ε, έχουμε τη βάση για την επόμενη προγραμματική περίοδο που θα είναι αυτός ο κανονισμός. Θα πρέπει να προσέξουμε να μην μειωθούν οι δυνατότητες συνεργασίας αλλά να διευρυνθούν και τα μέσα, οι πόροι να μην περικοπούν, τουλάχιστον να διατηρηθούν όπως έχει. Και η γραφειοκρατία που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια να αποδομηθεί. Και άλλη πρόοδος του κανονισμού είναι ότι δεν περιορίζεται μόνο η συνεργασία στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά με τα μέσα της ε, πολιτικής γειτονίας και της αναπτυξιακής πολιτικής μπορεί να ε, συνδεθεί και να προχωρήσει προς τα εκεί. Ο συνάδελφος Πασκάλ Νταριμόντ βελτίωσε πάρα πολύ την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πραγματικά το ε, αξίζει αύριο υποστήριξη από μεγάλη πλειοψηφία. Ζητώ συγγνώμη, λέει στα πολωνικά ο μιλητής ε, που υπερεύει το χρόνο μου. Αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και αξίζει να αφιερώσουμε το χρόνο που του αρμόζει. Ευχαριστώ πολύ. Ο ε, Πρόεδρος, συμφωνώ ε, με την άποψή σας. Παρ' όλα αυτά, αμένα μου έπεσε ο κλήρος τώρα εδώ για να τηρώ το χρόνο μας. Ο κύριος Χέτσμαν. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κυρία Επίτροπε, Κύριε Πρόεδρε, το Interreg έχει μεγάλη σημασία γιατί άρρητα τα ενδοκινοτικά σύνορα και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Χαίρομαι λοιπόν γιατί επιβεβαιώθηκε η αξία αυτού του μέσου με ένα ξεχωριστό κανονισμό. Μιλάμε για απλούστευση, για ε, απλούστευση του κόστους, χαμηλότερα, χαμηλότερο άχθος και διαχείριση εκ του σύνεγγης, ε, καθώς και συγκεκριμένα καταποκοπήν ποσά. Η διασυνοριακή συνεργασία ε, είναι πολύ μεγάλη σημασίας και αντικατοπτρίζεται και δημοσιονομικά. Ελπίζω λοιπόν να γίνει πλήρης χρήση του μέσου αυτού εδαφικής συνεργασίας. Μιλάμε για μια οροφή 85% για τη συγχρηματοδότηση, την οποία, η οποία βρίσκει σύμφωνο επίσης το 1 συν 3 μετατοπίζεται στο 1 συν 2, αλλά δυστυχώς πολλές φορές δεν υπάρχει χρόνος για τη χρήση των κατάλληλων πόρων. Συμφωνώ με αυτά που είπε και ο κύριος Ζέλερ μόλις πριν. Ναι, συμφωνώ και με τον κύριο Ζέλερ και σας ευχαριστώ που τηρήσατε το χρόνο σας. Βαλκάρσελ Σίζο, αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Παρά το γεγονός ε, ότι υπάρχει μία κλειστή λογική που χρησιμοποιείται, αυτό που έχει σημασία είναι η ευημερία των πολιτών και αυτό γίνεται προοδευτικά. Αυτό το βλέπουμε και στην Ισπανία και Πορτογαλία, διότι μετά το 89 η συνεργασία της διοίκησης βοήθησε το Αλεντέσου, το Αλκάρβε, την ε, Γαλλικία και αυτό μέσω του Ιντερεκ που αποτελεί μία όμορη γραμμή συνεργασίας η οποία βοηθά και Πορτογάλους και Ισπανούς. Έτσι υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στα σύνορα και ελπίζω να μην γίνουν περικοπές στο επόμενο πολιετές. Η πολιτική συνοχής θα πρέπει να δώσει μια νέα ε, όθηση στα σχέδια αυτά. Παρά το γεγονός ότι αυξάνεται ο λαϊκισμός, θεωρώ ότι μπορούμε να φτιάξουμε οδικά δίκτυα και να βελτιώσουμε την εκπαίδευση. Θέλουμε να άρουμε τα προσκόμματα και γι' αυτό είμαστε υπέρ της ε, ειρηνικής συνύπαρξης για μια περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη και ξεκινούμε από το Interreg. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα περνάμε στο Catch the Eye. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ζητήσατε το λόγο μόνο εσείς όσοι δεν είχατε λάβει το λόγο πριν. Ο κύριος Μπούντα, η εδαφική συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει μεγάλη σημασία για τη βελτίωση συνεργασίας των περιφερειών. Φτάσαμε σε αυτά αποτελέσματα ως προς την χρηματοδότηση που έγινε μέσω Interreg. Θεωρώ όμως ότι θα πρέπει να υπάρχει ενισχυμένο management σε περιφερικό επίπεδο για να έχουμε ομαδοποίηση συνεργασίας. Θα πρέπει να μιλάμε για οργανώσεις ενίσχυσης και περιφερειακής ενσωμάτωσης με βάση ένα κοινό στόχο α, περιφερειακής ανάπτυξης. Με αυτή την έννοια δέχομαι την συνεργασία δημάρχων της Ρωμανίας που δημιούργησαν τη Συμμαχία της Δύσης μέσα στα πλαίσια της περιφερειακής συνεργασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Νταμάτο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη δουλειά που έχει γίνει. Η αρχική πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αρκετά σημεία στα οποία είχαμε σταθεί επικριτικά και άλλωστε τροποποιήσαμε μέσα από τις συνομιλίες ε, είναι πολύ σημαντικό να υποστηριχθούν και τα θαλάσσια διαπεριφερειακά ε, προγράμματα που ενισχύουν ιδιαίτερα τη διασυνοριακή διάσταση. 11 δισεκατομμύρια σχεδόν χρειάζεται να είναι η οικοδότηση του Interreg με χρηματοδότηση 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή με προχρηματοδότηση. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές έτσι θα έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτούν τα έργα τα οποία αναπτύσσονται στην περιοχή τους, οι συναδελφοί οι οποίοι θέλουν να, παρα, να τροποποιήσουν τις παράλογες ε, διατάξεις της ε, οικονομικής διαχείρισης καλούνται να υποστηρίξουν τις προτάσεις μας για την έκπτωση των υπολογισμών και για την εθνική χρηματοδότηση. Έτσι λοιπόν μπορούμε να δούμε πραγματικά ποιος είναι υπέρ της ανανέωσης στην Ευρώπη και ποιος κατά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και για την συντομία στο χρόνο. Η Επιτροπός έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ιδιαίτερα κύριε Σιγητά, άκουσα με προσοχή τη συζήτηση και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω πως εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Ευρωπαϊκή Δαφική Συνεργασία παραμένει ουσιώδες στοιχείο της ε, ε, πολιτικής της συνοχής, της ευρωπαϊκής πολιτικής. Ακούσαμε με προσοχή τις απόψεις που εκφράστηκαν κατά τη συζήτηση. Ιδιαίτερα θέλω να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξη που προσφέρετε στην ε, ανάπτυξη των καινοτόμων επενδύσεων. Η Επιτροπή πιστεύει και εκείνη από την πλευρά της ότι με βάση την εμπειρία που είχαμε και από το παρελθόν θα υπάρξει μεγάλη ζήτηση για τους πόρους αυτούς. Αγαπητοί κυρίε και κύριοι βουλευτές, έχει γίνει καλή δουλειά μέχρι τώρα. Τώρα πια θέλουμε να εξασφαλίσουμε πως θα έχουμε ένα πιο απλό, αποτελεσματικό πλαίσιο για το μέλλον. Είμαστε βέβαιοι πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα σταθεί ισχυρό σύμμαχο στο πλευρό μας στο έργο αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω και ελπίζω, είμαι αισιόδοξη ότι τη Ρουμανική Προεδρία θα καταστεί δυνατό και για το Συμβούλιο να εγκρίνει στο δικό του κομμάτι τι προτάσεις Interreg προκειμένου αυτές ε, να ε, υιοθετηθούν μέσα στο 2019 πριν να ξεκινήσει ο προσεχής προγραμματικός κύκλος και ξέρετε φαντάζομαι όλοι πόσο σημαντικό είναι και αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ που έχετε μένει εδώ μέχρι αυτή την προχωρημένη ώρα. Και καλή σας νύχτα. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ και εγώ την Επίτροπο που έμεινε εδώ και που υπομονητικά παρακολουθεί τη συζητήση μέχρι το τέλος και δίνω το λόγο στον κύριο Άρημον, τον εισηγητή. Πρόεδρε, έχω εγώ την τιμή να ε, χρησιμοποιήσω τα δύο τελευταία λεπτά αυτής της κοινοβουλευτικής μας ημέρας. Δύο λεπτά τα οποία δεν θα μου αρκούσαν για να πω παρά μόνο να ευχαριστώ τους, τους συναδέλφους που συμπαραστάθηκαν στην ε, δουλειά αυτή, τους σκιώδης ε, που ήταν σε όλες τις συνεδριές των σκιωδών και που με πολλή δουλειά βοήθησαν να σταθεί ένα κείμενο ε, πολύ καλό και λογικό. Ένα ευχαριστώ για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που παρακολούθησε πάντοτε και στάθηκε στο πλευρό μας τη διαδικασία αυτή και θα ήθελα ολοκληρώνοντας να δείτε πόσο και την ε, παράκληση η Ρουμανική Προεδρία να δείξει τέτοια ε, προθυμία και να ετοιμάσει το general approach το ταχύτερο δυνατό ώστε να περάσουμε στον τριμερή διάλογο και να επιχειρήσουμε στο μέγιστο δυνατό να επεξεργαστούμε όλα τα στοιχεία του κειμένου πριν περάσει η σκητάλη στο προσεχές κοινοβούλιο. Ε, πιστεύω ότι είναι σαφές το κείμενο ε, εν ώψη της προσεχούς προγραμματικής περίοδου ε, προσφέρει δηλαδή ένα κείμενο το οποίο επιτρέπει στους ε, δραστηριοποιημένους στον τομέα αυτών όλα τα εργαλεία για να μπορέσουν να ετοιμαστούν και πάλι ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία και ελπίζω ότι θα συνεχίσει το ε, και στο μέλλον ισχυρό. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ τον εισηγητή, λέει ο Πρόεδρος. Εδώ ολοκληρώνεται η συζήτηση. Θα συνεχίσουμε αύριο Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου, από τις 8.30 έως τις 12.30 και από τις 3 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα. Τα πρακτικά δημοσιεύονται στον ιστοτοπό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πριν κλείσω για άλλη μια φορά ευχαριστώ την Επίτροπο.